Okay, friends, uh, Σας παρακαλώ. And see to that you have your voting cards. Ετοιμαστείτε παρακαλώ για την ψηφοφορία κυρίες και κύριοι να πάρετε και τις κάρτες σας, βάλτε τις στην προβλεπόμενη σχισμή στα έδρανά σας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Επαναλαμβάνω παρακαλώ τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Okay, Φίλες και φίλοι, αν είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία για την απόσπαση εργαζομένων στα πλαίσια της πρόσφορας υπηρεσιών με εισηγήτρια την κυρία Μωράν Σαρτιέ και την κυρία Ιονγκέριους. Ας αρχίσουμε με... Θα αρχίσω με την εξής ανακοίνωση. Η συμβαστική τροπολογία ε θα γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Εάν, εάν 11 μέλη, 11 μέλη το υποστήριξουν. Δεν έχουμε όμως φτάσει ακόμη εκεί. Ας αρχίσουμε με τη συμβαστική Β, B. Παρακαλώ ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει η τροπολογία 257. Ερχόμαστε στην 258, την οποία ψηφίζουμε μαζί με την 25 της ΣΥΜΚΟ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κάποιος ζητά επαλήθευση 258 μαζί με την 25 της ΙΜΚΟ. Δύο ψήφοι παραπάνω ε, σημειώνονται εδώ, μία παραπάνω για το Λαϊκό Κόμμα. Εντάξει τώρα, μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Εδώ λοιπόν κλείνει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ απορρίπτεται 34 κατά 259 αυτή όμως έχει αποσυρθεί τροπολογία 260 εκπίπτει όχι δε, η πρόεδρος την ψηφίζουμε την 260 τροπολογία 260 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωρώ. 262 τροπολογία αυτή εκπίπτει. Δεν έχω ακόμα συνηθίσει την ε, λίστα ψηφοφορίας ε, σε λίγα λεπτά. 262 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία συμβαστική F αυτή δηλαδή υπέρ κατά αποχές Παρακαλώ να επαναλάβουμε συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 275 μαζί με την 343 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Γιούρι 29 υπέρ κατά αποχές Νομίζω, μάλλον να επαληθεύσουμε λέει ο Πρόεδρος. Γιούρι 29, αρχίζει η ψηφοφορία. Μία πλεονάζουσα ψήφος σημειώνω στο, σημειώνεται στο Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. Οι 276, 277, 80, το και συνεχίζω μερικές σελίδες μέχρι τη σελίδα 12 όλες αυτές εκπίπτουν τώρα η 311 σελίδα 12 αρχίζει η ψηφοφορία α όχι με συγχωρείτε σηκώστε τα χέρια σας ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στη σελίδα 17, 349 τροπολογία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, όχι απορρίπτεται, συγγνώμη, 351 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. Συμβαστική age. ήτα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σί γάμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 38. Συμβαστική D, Δέλτα. Σελίδα 38. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί σελίδα 49 συμβαστική α λέει η πρόεδρος σελίδα 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σελίδα 51 51 λοιπόν, συμβαστική ε, ονομαστική ψηφοφορία έχει ζητηθεί. Υπέρ, ποιος είναι υπέρ της ονομαστικής ψηφοφορίας παρακαλώ να ηγερθεί. Άρα, ονομαστική ψηφοφορία για την συμβαστική ε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας για την ε, ε και προχωρώ σελίδα 52 τροπολογία 490 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική ε, G στη σελίδα 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 55 5, τροπολογία 500. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 13, νομικής επιτροπής, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σελίδα 57, συμβαστική Y, Y δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 58, συμβαστική Y, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 59, τροπολογία 520 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σελίδα 60. Προφορική τροπολογία. Έχετε σχόλια. Έχετε ενστάσεις μάλλον. Ο, μάλιστα δεν ψηφίζουμε λοιπόν λόγω του μεγάλου ρυθμού των ενστάσεων. Προχωρώ συμβαστική J υπέρ εγκρίνεται λέει πρόεδρος τώρα κατά όμως αποχές εγκρίνεται Α, να επαληθεύσουμε την συμβαστική J. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψηφί υπέρ. Προχωρώ στην σελίδα 61, τροπολογία 36. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και αυτή. 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L, λάμδα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωρώ στην συμβαστική μη. Σε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε 65 συμβαστική εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 66, Γιούρι 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Αυτή εκπίπτει. Συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 70, συμβαστική Q, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 72, τροπολογία, ΙΜΚΟ 10, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 102 μαζί με την 103 Α, αυτή έχει αποσυρθεί όμως 102 μόνο λοιπόν τίθεται σε ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική σίγμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 76. Αρχίζομαι με... με τη συμβαστική ΤΑΦ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική X, σε 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 79 συμβαστική κάπα υπέρ. Κάπα λοιπόν, 79 σελίδα. Η 143 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική κάπα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 83. Συμβαστική, συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, U μάλλον, U. Σελίδα 85, συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση, όπως κατάλαβα, για την συμβαστική τροπολογία V. V, όπως Victory, αρχίζει. Τώρα πέρας εγκρίνεται υπέρ 38 ψήφι. Ε, συνεχίζομαι. Σελίδα 88. Ήμκο 20. Καθώς και η υπαριθμόν 200 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Σελίδα 89, τροπολογία 203, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 93, συμβαστική Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 224. Α, με συγχωρείτε αυτή η εκπίπτη. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται. Επαλήθευση. Καλώς. 225 επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και πέρας τώρα. απερίφθη με μικρή διαφορά μιας ψήφου. Συμβαστική ΑΑ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΑΒ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 97, προγείο 244, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε όμως τον 244. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψήφι 35 υπέρ, 16 κατά. 246 υπέρ, κατά. Αποχές Επαναλαμβάνουμε τη 246 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 253 έχει αποσυρθεί. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία αυτή τη φορά. Άρχισε τώρα. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ και όλες εννοείται την τελευταία αυτή ψηφοφορία. Μάλιστα. Ε, πέρα της ψηφοφορίας. Ε, ενεκρίθη. 32 ψήφοι υπέρ. 8 ψήφοι κατά και 13 άποχες. Τώρα, πρέπει να ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Χρειάζεται το λιγότερο 28 ψήφοι υπέρ για να εγκριθεί η διαπραγματευτική εντολή. Αρχίζει η ψηφοφορία λοιπόν τώρα, όπως είπα, εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Και Τέλος. Ω, βλέπω ότι είναι μια ισχυρή εντολή, εντολή με 44 ψήφους υπέρ και 8 ψήφους κατά. Ε, συγχωρείτε. Να με συγχωρείτε κυρία Σάρτχε θα σας δώσω το λόγο σύντομα, αλλά, λέει ο πρόεδρος Ουλφσκογκ, έχω την κυρία Λαμπάτζοβα που επιθυμεί να καταθέσει δήλωση εκ μέρους της μειοψηφίας. Α, εσείς κύριε Μαρτά. Δήλωση εκ μέρους της μειοψηφίας. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό κύριε. Κυρία Πρόεδρε, θα βρείτε τις αιτιολογικές σκέψεις μας εντός του εγγράφου. Η ομάδα μας, Ευρώπη των Εθνών και Ελευθεριών, δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εργασία που εκφράζει η έκθεση. Αναγνωρίζουμε κάποιες προσπάθειες για την σκρίνηση της νομοθεσίας. Θεωρούμε όμως ότι το κείμενο δεν κινείται επαρκώς μακράν και γι' αυτό δεν επιθυμούμε να το ενισχύσουμε. Κύριε Αλαμπάντζοβα, δεν είχατε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχα αντιληφθεί ότι πρέπει να το πράξω και προφορικός, νόμιζα μόνο γραπτός. Εγώ ψηφίζα μόνο για ίδιο λογαριασμό. Θεωρώ ότι η ισορροπία μεταξύ ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και προστασίας των εργαζομένων δεν εξασφαλίζεται και γι' αυτό ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Η πρόεδρος Ουλφσκοκ χωρί μικρόφωνο. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μωράν Σαρτιέ, συνεισηγήτρια. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ που προεδρέσατε τέλεια εδώ, αλλά θα έπρεπε να σκεφτώ και τον Τόμα Χέντελ, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, δεδομένως τη σημασία αυτού του κειμένου για την κοινωνική Ευρώπη, για αυτή τη νέα οδηγία, για τη σημασία των όσων έκανε η Επιτροπή απασχόληση τη εργασία του Κοινοβουλίου για μια νέα Ευρώπη πιο κοντινή στους πολίτε, Βεβαίω θα έπρεπε να είναι εδώ ε, και πραγματικά το σκέφτομαι σήμερα. Να ευχαριστήσω και το Γιάννης ε, Ιουγγέριους με τον οποίο συνεργάστηκα πολύ στενά ε, ε, να ευχαριστήσω τους πολιτικούς μας συμβόλους, τους βοηθούς μου ούτε και ξέρω πια ποιος έκανε τι σε αυτή την τόσο πλήρη ομάδα εργασίας και βεβαίως θα ήθελα να εκφράσω μια σκέψη και μια ευχαρίστηση προς τους, ε, μια ευχαριστία προς τους σκιώδεις γιατί είχαμε 18 μήνες σκληρή δουλειά για μια πραγματική ε, κοινωνική Ευρώπη, μια ισορροπία για τους μισθωτούς ολόκληρη την Ευρώπη και ισορροπία για τις επιχειρήσεις. Είμαι πολύ περήφανη για αυτή την εργασία ε, και ευγνώμων στο σύνολο της Επιτροπής Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν να χάσω τελείω τη φωνή μου σήμερα να πω ότι δύο πολύ δυνατές γυναίκες, δύο ισχυρές γυναίκες είναι φανταστικό το σημερινό. Ευχαριστώ όλους. Next meeting in the committee. Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 19 Οκτωβρίου 9 με 12 εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Αντίο